E, Άρχεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά τη τελευταία συνεδρίαση είναι διαθέσιμα. Μήπω υπάρχουν παρατηρήσει για τα πρακτικά. Όχι. Οπότε εγκρίνονται πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ώρα των ερωτήσεων προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Θα ήθελα να, να καλωσορίσω τον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, ο οποίος έρχεται εδώ κάθε μήνα για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι κανονισμοί είναι ίδιοι, οι κανόνες είναι ίδιοι. Ένα λεπτό για την ερώτηση, ένα λεπτό για την απάντηση, δεν έχουν αλλάξει και ενδεχομένως υπάρχει δυνατότητα ε, ε, να δοθούν 30 συμπληρωματικά δευτερόλεπτα για την απάντηση, μια συμπληρωματική απάντηση αν το κρίνει σκόπιμο πρόεδρος. Για το ΕΛΚ. Ο κύριος Ιωάννης Χασουλίδης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Μπαρόσο, εξ ονόματος του Προέδρου Ντόλ, Θέλω να σας υποβάλω το εξή ερώτημα. Η ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελε να γνωρίζει τις απόψεις σας σχετικά με τις τωρινές προσπάθειες για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Παλαιστινιακού θέματος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες τους να πείσουν το Ισραήλ να παρατείνει το δικαιοστάσιο για την επικισμό στην Δυτική Ιερουσαλήμ και την Λωρίδα της Γάζα δεν οδηγούν πουθενά οι προσπάθειες να αναλυφθούν χωριστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κουαρτέτο για να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις εν ώψη των εξελίξεων πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε την επανάληψη της προθυμίας Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος όποτε αυτό θα είναι εφικτό και κατάλληλο. Ποια είναι η εξολόγησή σας για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Ρωρίδα της Γάζας μετά την απόφαση του Ισραήλ το 2010 να διευκολύνει την κυκλοφορία και να καταλάβει προσπά... καταβάλει προσπάθειες για την απελευθέρωση Thank As you know, the European Union... την απελευθέρωση των, διαδρόμων. Είμαστε υπέρ τη επανάληψη των συζητήσεων και των συνομιλιών. Ο πρόεδρο του Συμβουλίου παρουσίασε χθε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να δεχθεί νέο πάγωμα το, του επικισμού το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Η κατάσταση μα απογοήτευσε κυρίω επειδή δημιουργεί των κατάλληλων συνθήκων για μια λύση δύο κρατών δεν είναι κάτι που θα ωφελήσει την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό τη, αλλά είναι και προ το συμφέρον του Ισραήλ κατά την άποψή μου. Για τι διαπραγματεύσει, το ε, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών αποφάσισε να, την παρέμβαση του Κουαρτέτο, ειδικό ε, εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συναντήσει την κυρία Άφσον για να την ενημερώσει για τι τρέχουσε, τι πρόσφατε εξελίξει. Στηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή και το Κουαρτέτο θα μπορούσε να, να ε, επαναλάβει τι δραστηριότητέ του. Η κυρία Άστον είναι σε επαφή με εκπροσώπου της περιοχής και θα είμαστε παρόντες στη συνεδρίαση του Συμφώνου των Αραβικών Κρατών διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε σαν λύση το αδιέξοδο. Ε, πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με τις ΗΠΑ θα βρεθεί μια λύση. Yes, Συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω και πάλι σχετικά με την ανθρωπική ανθρωπιστική κατάσταση της Λωρίδα της Γάζας μετά το άνοιγμα των διαδρόμων και τι συμβαίνει με τον Τζιλάλ Σαλίντ η οικονομική ανάκαμψη απαιτείται απαραίτητο, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει πολιτική στη Γάζα την οποία ζητάμε τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα να υποστηρίξει ε, τους εμπειρογνώμονες μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού Φαγιάντ. Εγώ δέχθηκα τον Πρωθυπουργό Φαγιάντ και είχαμε συνομιλίες για το θέμα αυτό, διότι πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ο κύριος Σούλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαρόζο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν εάν έχετε την άποψη ότι η θέσπιση των εισαγωγή των ευρωομολόγων για την σταθεροποίηση του ευρώ μπορεί να συμβάλλει θετικά. Δεύτερον, συμμερίζεστε την άποψη τη ε, κυρία Άγγελα Μέρκελ, τη Γερμανίδα Καγκελαρίου, ότι τα ευρωομόλογα δεν είναι αναγκαία. Τρίτον, τι θεωρείτε για την περίπτωση που έχετε διαφορετική άποψη από την κυρία Μέρκελ, εάν είστε υπέρ δηλαδή των ευρωομολόγων, τι σκέφτεστε να κάνετε την προσεχή Πέμπτη στο Συμβούλιο. Πέμπτον, συμφωνείτε με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Juncker, Είστε σε επαφή μαζί του και θα τον υποστηρίξετε. Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην περίπτωση που δεν θα προχωρήσετε σε ευρωομόλογα, ε, πώς θα αντιδράσετε σε αυτή την απόφαση της μη έκδοσης ευρωομολόγων. Ε, η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο αυτό ήδη το 2008 στο έγγραφό της αλλά ωστόσο εντωμεταξύ θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση ε, δημιούργησε το SMF και αυτά τα εργαλεία δεν, είναι, δεν έχουν ένα εξαντλητικό χαρακτήρα αλλά μπορούν να, θα πρέπει να βελτιωθούν για να είναι πιο αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε το απλό ερώτημα. Αντιμετωπίζουμε καλά την κρίση μέσω συνενετικών εργαλείων ή μέσω ε, τρόπων που ενδεχομένω είναι πιο αποτελεσματικά αλλά δεν τη χάνουν γενική συνένεση. Και όπω είπατε δεν υπάρχει συνένεση όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Γιούγκερ. Άρα λοιπόν η απάντηση σήμερα είναι προφανής. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε εργαλεία που μπορούν να τύχουν συνένεση στην Ευρωζώνη. Γιατί αλλιώς αυτό θα είναι ει βάρο της ε, αγοράς. Λοιπόν, ας μην ε, αποκλείσουμε την ιδέα των ευρωομολόγων για το μέλλον, αλλά σε επικεντρώσουμε την προσοχή μας αυτή τη στιγμή σε αυτό που μπορεί να λειτουργήσει τάχιστα και αποφασιστικά. Ναι, ε, απαντήσατε διπλωματικά κύριε Μπαρόζο, αλλά δεν θα ήθελα να το αφήσω να περάσει. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω μια ακριβέστερη ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός ο κύριος Γιούγκερ στην λειτουργία του ως ο πρόεδρος του Ευρωγκρουπ εξήγηλε ότι πρόκειται να υποβάλει μια πρωτοβουλία στο Συμβούλιο για την εισαγωγή των ευρωμολόγων. Θα τον υποστηρίξετε και ενδεχομένως θα προσπαθήσετε να πείσετε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή να προσχωρήσουν στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών ή θα πείτε στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σαρκοζή ότι εντάξει, συμφωνούμε μαζί σας και υποχωρούμε. Ε, δεν ε, πιστεύω ότι υπάρχει ελάχιστη ε, δυνατότητα αυτή τη φάση να πετύχουμε μια συμφωνία για τα ευρωμόλογα. Υπάρχει προθυμία εκ μέρου πολλών χωρών μελών όσον αφορά αυτή την πρόταση. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την πλατύτερη δυνατή συνένεση με τα υπάρχοντα εργαλεία. Σα είπα ειλικρινά, κύριε Σούλτ, ότι θεωρώ ότι η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, ελκυστική και πράγματι. επίτροψά έκανε κάποιες ε, ε, έχουν υποβληθεί κάποιες ε, προτάσεις από, διαφόρους, ε, από εξαιρετικούς προκατόχους μου σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο, κύρι... Ο κύριος Φερχόφστατ, μια συγκεκριμένη ερώτηση κύριε Μπαρόσο. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία. Μπορείτε να προχωρήσετε με μια πρόταση για τα ευρωμόλογα. Αυτή ήταν η ερώτηση που έθεσε ο κύριο Σόλτ. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό προ το παρόν. Έχω συγκεκριμένη ερώτηση για την απαλλαγή του 2009. Υπάρχει μια βεβαίωση, ε, δήλωση διαβεβαίωση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής που αναφέρει ότι 38 από τα 39 προγράμματα η Γενική Διεύθυνση δεν έχει επαρκή ε, διαβεβαίωση για την νομιμότητα και, την, ε, το σωστό τρόπο των καταβολών των δηλώσεων που έχουν δηλωθεί για, των δαπανών που έχουν δηλωθεί για το 2009. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε αυτή την ε, βεβαιότητα και η δήλωση συνεχίζει. Ε, για τα υπόλοιπα 41 προγράμματα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε φάση πρώτερη πριν το 2009. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Εφόσον αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη των δηλώσεων αυτών, τι πολιτική, τι δράση θα αναλάβετε έναντι των κρατών μερών. Καταρχά, κύριε Φεχόφστα, να σα πω ότι το δικαίωμα πρωτοβουλία τη το έχει ήδη χρησιμοποιήσει η Επιτροπή. Όταν ξεκίνησε ο μηχανισμό, ο κύριο Ρεν και εγώ είχαμε προστρινή μια δυνατότητα συλλογικών εγγύσεων που πήγαινε προ την κατεύθυνση των ευρωομολόγων το οποίο απερίφθη ρητά από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να έρθουμε μια, με μια νέα ε, ε, πρόταση που θα διαιρεί και πάλι τα κράτη-μέλη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Υποβάλλουμε επίσημα προτάσει όταν. Ε, ε, η λύση όταν γίνονται αποδεκτές. Δεν υποβάλλουμε όταν υπάρχει μια κατάσταση διχόνοια στο εσωτερικό των κρατών μελών. Οι προτάσεις αυτές υποβλήθηκαν από την Επιτροπή και απορρίφθηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για τις δημοσιονομικές προοπτικές ήδη δεσμεύτηκα να υπάρξει πρόταση συγκεκριμένου είδους ευρωομολόγων για ευρωπαϊκά έργα και ήδη έλαβα νητικά σχόλια από κάποιες ε, πρωτεύουσες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να ελπίζω ότι θα γίνει. Για την ερώτησή σας και συγγνώμη απάντησα στο σχόλιο που κάνετε. Για την ερώτησή σας θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα από τα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, με κάποιες εξαιρέσεις 4-5 κράτη, τα περισσότερα δεν μπορούν να δώσουν αυτή τη ε, δήλωση διαβεβαίωση. Είπατε, σωστά είπε η Γενική Διεύθυνση που αναφέρεται ε, αυτά που είπε και έχουμε όλα τα εργαλεία για να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εμπλακούν όσο νωρίτερα γίνεται στον έλεγχο της δαπάνης των κοινωτικών κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο Μποβέ. Κύριε Μπαρόσο, πριν από ένα χρόνο μας είχατε πει στη διάρκεια της πρώτης εντολής ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είχαν δηλητηριάσει την εντολή σας και θέλετε να παραπέμψετε το θέμα στα κράτη. Πριν από λίγες μέρες συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές ε, υπογραφές για μια πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητη για τους ε, οργανισμούς αυτούς. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και Γεωργίας ε, απέριψε την πρόταση του Επιτρόπου Ντάλι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έδωσε αρνητική ε, γνώμη. Έχουμε και το σκάνδαλο στην ΕΦΣΑ και τα θέματα που έθεσε το πάνελ. Η ΕΦΣΑ ήδη αποφάσισε να ε, δημοσιεύσει νέες κατευθυντήρες γραμμές αξιολόγησης. Είστε διατεθειμένος απόψε να δεχθείτε οποιαδήποτε ανανέωση καθό, όσο οι νέοι κανόνες που θα εφαρμοστούν από την ΕΦΣΑ δεν θα έχουν εγκριθεί. Η νέα αξιολόγηση και η νέα διαδικασία διοδότησης πρέπει να ακολουθεί, να γίνει με βάση τους νέους κανόνες. Είστε διατεθειμένος να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ώστε να έχουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Κύριε Μπουβέ, σας ευχαριστώ. Πέρασε ο χρόνος σας. Σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή, όπως ξέρετε, δεν ισχύει ακόμα αυτό το νέο καθεστώς. Και βεβαίως παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες των πολιτών για αυτό το θέμα. Ο αρμόδιος επίτροπος ε, παρακολουθεί και αυτός ε, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες παρόλο που επίσημα δεν έχουμε εγκρίνει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Σε ό,τι αφορά το θέμα θα εξακολουθεί να ισχύει η τρέχουσα νομοθεσία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η ΕΦΣΕ είναι μια, ένας ανεξάρτητος οργανισμός γνωμοδοτικός και πρέπει βεβαίως να σεβόμαστε τις απόψεις, τις γνώμες αυτού του ανεξάρτητου οργανισμού. Θα σε, να σεβόμαστε και να τηρούμε σε αυτό το θέμα το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούμε να αναστείλουμε την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε επιτροπή. Δεν με ικανοποιεί το καθεστώς των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δεν είναι απόλυτα σαφέ, αλλά είναι το μόνο καθεστώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι υποχρεωμένο να το τηρώ. Once again, Mr. και πάλι. Η απάντησή σας... Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά υπάρχουν νέε κατευθυντήρε γραμμές, τις οποίες καθιέρωσε η ΕΦΣΤΑ, που είναι πολύ πιο αυστηρέ. Όλε οι νέε άδειε που χορηγήθηκαν ε, πρόσφατα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση τις νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αξιολογήσει σήμερα με βάση παλαιών κανόνων, προηγούμενων κανόνων. Θα ήθελα λοιπόν να λύσετε αυτό το θέμα και να ξαναρχίσετε αυτή τη συζήτηση η οποία πρόκειται να γίνει το 2012. Η επικαιροποίηση της οδηγίας ε, είναι μια διαδικασία που πρέπει να προχωρήσει. Όπως πάντα λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις και τις υποδείξεις της του ανεξάρτητου οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων, της ΕΦΣΑ. Και αν μα προτείνει νέε κατευθυντήρε γραμμέ, θα τι μελετήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Το μόνο που μπορώ να σα πω τώρα είναι αυτό. Αλλά το νομικό καθεστώ για την έγκριση για των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα εξακολουθεί να ισχύει αυτή τη στιγμή εκτός αν κάτι αλλάξει. Πάντως με πολύ μεγάλη προσοχή θα μελετήσουν αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμίνσκι, πρόεδρος του ΙΣΕΡ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε Μπαρόζο, από τις 19 Απριλίου η Gazprom και το Consortium Nord Stream κατασκευάζουν αυτό το μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου. Δεν θα μιλήσω πάλι για τις περιβαλλοντικές ε, διαστάσεις του έργου αυτού, γιατί τις συζητήσαμε ήδη. Εφιστώ την προσοχή σας στο εξή, διότι μπαίνουν οι σωλήνες αυτή την εποχή, που ενοχλούν την είσοδο των ε, μεγάλων σκαφών σε ένα πολωνικό λιμάνι που δημιουργεί, που παράγει θέσεις εργασία ε, για πολλούς Πολωνούς στην Ανατολική Πολωνία. Μερικοί από αυτού έχασαν τη δουλειά τους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εμείς το θέσαμε διμερώς το θέμα ω Πολωνία, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού. Διότι ε, από την άλλη μεριά των συνόρων ε, κοντά στο Στετίνο υπάρχει το λιμάνι του Ροστόκ και προσπαθούν να προωθήσουν το Ροστόκ. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια θα πρέπει να είναι ισότιμα σε επίπεδο ανταγωνισμού και να μην ενοχλεί ένα λιμάνι του ότι γίνεται σε άλλο κράτος μέλος. Γνωρίζω ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποια από αυτά τα λιμάνια που αναθέσετε. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ε, η γερμανική αρμόδια υπηρεσία ζήτησε από την Northrim να, να προετοιμάσει ένα αναθεωρημένο, μια αναθεωρημένο σχέδιο για το τμήμα του αγωγού που περνάει από το, κοντά από το πολωνικό έδαφος και από τα χωρικά είδατα της Πολωνίας για να μην υπάρξει παρεμνόχληση ε, των λιμένων. Ως αποτέλεσμα θα κάθονται, τα ισολίνε αυτοί θα απέχουν ε, σε 20 ή 20 χιλιόμετρα από τις ακτές ε, πάνω στον πυθμένα της θάλασσας. Επιπλέον, ε, ο πρόγραμμα, η, η αμφισβήτηση σχετικά με το, τη διαδρομή του, του αγωγού οδήγησε σε μία απομάκρυνση του αγωγού από τις ακτές 12 χιλιόμετρα. Οι γερμανικές αρχές και, και ο ανάδοχος έχουν αναλάβει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες τόσο ώστε κάθε περιορισμός πρόσβασης σε πολωνικούς λιμένες να, ε, να μην δημιουργεί κανένα πλέον πρόβλημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε ισότιμα τα κρατη Θα ήλπιζα ωστόσο ότι αυτή τη φορά η Επιτροπή ε, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία ισότιμα πραγματικά. Πήρατε στοιχεία κυρίως από την Γερμανία. Ζητώ από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη και τα στοιχεία που παρέχει η Πολωνία. Μπορεί να στείλετε επιπλέον επιτόπου ανεξάρτητου ελεκτέ. Εγώ εμπιστεύομαι στην Επιτροπή ούτω ώστε να αντιμετωπίσει όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα κύριε Καμίνσκι. Όντω, εμεί παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στο ζήτημα αυτό και έχουμε επίγνωση του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματο και οικολογικά και από άλλες οπτικές γωνίες. Παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα με μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Μπίσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο. Αναφερθήκατε, απαντήσατε στο ερώτημα του κυρίου Σούλτς ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα πράγματα με τα ευρωομόλογα. Προηγουμένως ε, μας είπαν ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν πρόκειται να επιβληθεί και άλλα πράγματα, δεν, ε, άλλες προτάσεις δεν τελεσφόρησαν. Είμαστε, διανύουμε το τρίτο έτος μετά την έναρξη της κρίσης και ρωτώ ε, κατά πόσο θα ε, συμφωνήσετε με την προσπάθεια διάσωσης του ευρώ ή θα απορριφθούν πάρα πολλές προτάσεις τελικά το Σαββατοκύριο Σαββατοκύριακο. Το ερώτημα το οποίο θέτω είναι ποιο είναι το κόστος αυτών των, αυτής της διστακτικής τάσης εκ μέρου σας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε το εξή ε, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όταν ε, συναντιούνται, όταν συναντιόμαστε, γιατί και εμείς είμαστε μέλος του Συμβουλίου, δεν μιλούμε μεταξύ μας. Δεν είναι μας προς πολιτικούς, αλλά προς την αγορά. Άρα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν, θα πρέπει να κάνουμε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τα σχόλια τα οποία υποβάλλουμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και απάντησα πολύ ειλικρινά στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σούλτς διαπιστώνουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα πρόταση για τα ευρωομόλογα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να την αποκλείσουμε, να τη σκοτώσουμε, αλλά είναι προφανέ ότι υπάρχει συνένεση εκ μέρου των χωρών μελών. Και ε, δεν θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι το οποίο είναι προφανέ για μένα, αλλά διαιρεί τι χώρε μέλη. Ε, υπάρχουν ε, κάποιες συνενατικές λύσεις επί των οποίων μπορούμε να βασιστούμε ούτως ώστε να προστατεύσουμε το ευρώ και την ευρωζώνη. Σας ευχαριστούμε. Επιπρόσθετη ερώτηση εκ μέρους του κ. Μπίσκη, παρακαλώ. Κύριε Μπαρόζο, ένα σύντομο ερώτημα. Υπάρχουν άλλα εργαλεία τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί νομίζω ότι δεν είμαι καλά ενημερωμένος. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα εργαλεία για τα οποία συζητούμε θα πρέπει και να εφαρμοστούν απάντηση. Ε, συζητούμε πολλά, πολλές εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικά εργαλεία. Το τελευταίο Ευρωγκρουπ εξέτασε πολλές εναλλακτικές ε, δυνατότητες και διάφορες ιδέες και η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλα τα ενεχόμενα μέρη. Ε, εγώ ίδιος διαβουλεύομαι όχι μόνο με τις χώρες μέλη, αλλά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας, τον διευθυντή του ε, Νομισματικού Ταμείου κλπ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σόφρον όπως συνέβη ορισμένες φορές και το παρελθόν να κάνουμε μεγαλοσχήμονες εξαγγελίες που τελικά δεν εφαρμόζονται στην ε, πράξη. Νομίζω ότι αυτή τη φορά κάνουμε το αντίθετο. Θα καταλήξουμε σε κάποια από τα συμπεράσματα όταν είμαστε έτοιμοι. Και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεργάζεται με ενεργητικό τρόπο με όλες τις ε, χώρες ε, μέλη. Και θα δράσουμε όταν είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα. Ευχαριστούμε πολύ πρόσφατη θύλα των Wikileaks ε, δημιούργησε έντονα αισθήματα. Κάποιοι λένε ότι είναι καλή η διαφάνεια, άλλοι ότι δυσκολεύει τη διπλωματία. Μένα μου άρεσαν πολύ οι μνήε ε, στο Wikileaks ό,τι αφορούσε εσά. Όταν μιλούσε για το ταξίδι σα στη Ρωσία και το ότι αγνοήσατε και αποκλείσατε τη ρωσική άποψη ότι ήσασταν μόνο ένας έτσι αρκετά αναδεδειγμένο, δημόσιο, διεθνής δημόσιος υπάλληλο. Αυτό το έλεγα και εγώ σε εσά, Πρόεδρε. Σα είπα και σα ξαναείπα ότι δεν σα έχει εκλέξει ο λαό και για το λόγο αυτό δεν έχετε πραγματική νομιμοποίηση. Το γεγονό ότι δεν έχετε εκλεγεί είναι ο λόγο για τον οποίο δεν σε σέβονται περισσότερο διεθνώ και γιατί όλο ένα και περισσότερο οι λαοί της Ευρώπης θεωρούν ότι και εσεί και η Επιτροπή είσαστε άξιοι περιφρόνησης δεν πιστεύω ότι θα βρείτε, δεν περίμενω ότι θα είχατε κοινή άποψη με τους Ρώσους, αυτό λέτε εσείς, ε, προτείνετε, μάλλον λέτε ότι συμφωνείτε μαζί σας, μαζί τους. Να σας πω, εμένα με εξέλιξε το Κοινοβούλιο με μυστική ψηφοφορία. Άρα αξίζω την εμπιστοσύνη, αν μη τι άλλο και το σεβασμό, όλων των μελών του Κοινοβουλίου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει 27 δημοκρατίες και ο τρόπο εκλογής του Πρόεδρου τη Επιτροπή με τον τρόπο αυτό είναι εύλογο. Δεν είμαστε κράτο και δεν νομίζω ότι θέλετε να υπάρξει ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό κράτος. Εφόσον είμαστε λοιπόν ενωμένο κράτος, η άμεση εκλογή του, δεν υπάρχει άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής. Μπορεί να σας αρέσει, να μην σας αρέσει, εμένα μου αρέσει περισσότερο, αλλά εξελέγει από το Κοινοβούλιο υπάρχει ένας προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ορίστηκε από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Αυτός είναι ένα δημοκρατικός τρόπο αντιμετώπιση των διαφορετικών, τη Ένωση. Άλλοι δεν σέβονται τα θεσμικά όργανα τη Ένωση. Ήλπιζα τουλάχιστον ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου θα σεβόντουσαν του θεσμού της Ένωσης. Συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Μπαρόζο, μου άρεσε πάρα πολύ ε, το γεγονό ότι σήκωθήκατε και κομπάζετε διότι σας εξέλεξαν μυστικά και ότι αυτό θεωρείται πως σας δίνει νομ... δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό είναι το πιο απίθανο που έχω ακούσει σε όλη μου τη ζωή. Στην πραγματικότητα η Επιτροπή έχει το μόνο δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία που βλάπτει τις οικονομίες της Ένωσης και μόνο αυτή. Αν μήπως θα έπρεπε τα θέματα αυτά να το αποφασίσει ο λαός της Ευρώπης, οι λαοί της Ευρώπης με δημοψήφισμα. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ όλοι. Λυπούμε. Κύριε Σούλτς, κύριε Σούλτς, κύριε Σούλτς, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Συνάδελφοι, κοιτάξτε, κοινοβούλιο είμαστε. Κύριε Μπαρόζο οι εκλογές στο Κοινοβούλιο ήταν ανοιχτές. Και πολλοί θεωρούν ότι η, πιο ελεύθερη εκλογή είναι όταν ο κόσμος αποφασίζει μυστικά. Συνήθως τα ολοκληρωτικά συστήματα δεν επιτρέπουν μυστική ψηφοφορία ακριβώς για να αυξήσουν την πίεση στα άτομα. Πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα. τα περισσότερα πολιτικά συστήματα δέχονται και δημοψηφίσματα και αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και μάλιστα στη Βρετανία γεννήθηκε η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που είναι ένα εξαιρετικό τρόπο απόφαση στην δημοκρατία. Ε, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η κυριαρχία των κοινοβουλίων είναι βασική αρχή του κοινοβουλευτισμού. Η αντιπροσωπευτικότητα λοιπόν και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν μπορεί να λέτε ότι δεν εκπροσωπούν τη δημοκρατία, ότι δεν είναι δημοκρατικό μέσω έκφρασης των απόψεων. Ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Η Κίνα έχει μεγάλο πλεόνασμα στο εμπορικό της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παροχές υπηρεσιών είναι πάρα πολύ μικρές για να αντισταθμίσουν αυτή την κατάσταση. Το πλεόνασμα οφείλεται σε υποτίμηση του νομίσματος, σε με αποτέλεσμα οι εισαγωγέ να μην είναι δυνατέ, ενώ οι εξαγωγές γίνονται σε πολύ φθηνότερε τιμέ. Και αγνοεί τα, τα, τα, του κανονισμού που ισχύουν για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Η Κίνα συσσωρεύει από θέματα ξένου και ελέγχει τους ε, ε, ε, φυσικούς σπόρους του πλανήτη που έχουν αρχίσει να σπανίζουν. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό ανταγωνιστή που κινδυνεύει να καταστρέψει τη ζωή, μου, η Ευρω... τη ζωή μας. Οι ευρωπαϊκές χώρες μεμονωμένα συλλογικά πρέπει να προσθέσουν τη βιομηχανία τους. Γιατί η Επιτροπή επιτρέπει επιχειρήσεις και εργαζόμενους Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχονται τον αθέμητο ανταγωνισμό της Κίνας θα ήθελα να σας πω ότι θα είμαστε πιο επιτυχείς στις προσπαθειές μας αν τα ενεργήσουμε συλλογικά και όχι μεμονωμένα. Δηλαδή δεν μπορέσουμε να ασχίσουμε μεμονωμένα αρκετή πίεση για να εξασφαλίσουμε, εφαρμόσουμε κάποια μέτρα στην Κίνα. Συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει επαφέ με την Κίνα, αυτό το κάνουμε. Είμαστε υπέρ των ελευθέρων συναλλαγών, αλλά και υπέρ του θεμητού εμπορίου. Όταν υπάρχουν στοιχεία ενδείξει για ντάμπινγκ, εφαρμόζουμε κάποια μέτρα anti-dumping κατά της Κίνας. Δεν ήταν κάτι το εύκολο. Ορισμένα κράτη-μέλη είχαν αντίθετη άποψη. Το κάναμε παρόλα τα αυτά και συζητούμε Κάθε φορά που συναντούμε με την κινέζικη ηγεσία, συζητούμε το θέμα των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία και διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, ώστε να έχουμε ελεύθερε ανοιχτέ εμπορικέ σχέσει με αυτή τη χώρα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με στεναρότητα. Θέλουμε να πείσουμε την Κίνα για την υποχρέωσή τη να τηρεί ορισμένου κανόνε. Ευχαριστώ. Well, ερώτηση. Είπατε κύριε Μπαρόσο ότι πιστεύατε στο θεμητό εμπόριο. Το θεμητό εμπόριο δεν είναι αυτό που μας προσφέρεται. Αυτό που έχουμε είναι αθέμητο ανταγωνισμό, ε, αθέμητο εμπόριο υπέρ της Κίνας. Θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις για να ανατιμηθεί στο νόμισμα της ε, Κίνας. Θα ψεύεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνής που αποτελούν το 5% του ΑΕΠ της Κίνας. Μήπω η λύση θα ήταν να μπλοκάρουμε, να παρεμποδίσουμε τις ε, εισαγωγέ από την Κίνα το ζωθυμητό εμπόριο υποστηρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη, είμαστε υπέρ της αμοιβεβαιότητας. Αρχή της σημαίνει ότι θέλουμε να παραμένουν ανοιχτέ οι αγορέ και είναι προ το συμφέρον μα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, πιο σημαντικό και από την Κίνα. Είναι λοιπόν σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτέ οι αγορέ, αλλά οι εταίροι μα πρέπει να σέβονται ορισμένου βασικού κανόνε για τι συναλλαγματικέ ισοτιμίε στη συνεδρίαση του G20 θέσαμε αυτό το θέμα διότι πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσει όταν μιλάμε για τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία. Μπαίνουμε στο δεύτερο τμήμα με τη διαδικασία Catch the Eye και θέμα το Wikileaks και την κύβερνο ασφάλεια. Ο κύριος Καέλιο έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, δεν θα μιλήσω για την αμερικανική διπλωματία ή ε, τα υπέρ και τα κατά της πληροφορικής. Θέλω να σας μιλήσω για τον κύριο Ασάντζ. Υπάρχουν πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν και, ζητώ από, και ζήτησα από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών να επανεξετάσει την ε, ανάκριση που είχε ξεκινήσει το 2007 για τις δραστηριότητε της CIA στην Ευρώπη. Τότε η Επιτροπή Μπαρόζο, η προηγούμενη, στην προηγούμενη θητεία της, είχε συνεργαστεί και είχε βοηθήσει την προώθηση της διαφάνειας, αντίθετα από το Συμβούλιο που είχε πει ψέματα στο Κοινοβούλιο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Είναι η Επιτροπή σα πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, Πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, πάντα βοηθούσε με απόλυτη διαφάνεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν και θα το κάνει και στο μέλλον. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι λοιπόν, αυτό είναι λογικό και είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου να υπάρχει σεβασμός κριτηρίων και αρχών της διαφάνειας όσο αυστηρότερον γίνεται. Και βεβαίως τον θεσμικό διάλογο. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέρτσοκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα απλό ερώτημα. Οι Ευρωπαίοι είναι ουσιαστικά εξαρτημένοι ε, στις μέρες μας. Αλλά τα κριτήρια ασφάλειας για το ίντερνετ, τι γίνεται με αυτά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα για την Επιτροπή να υποβάλει κάποιες προτάσεις ε, για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης. Ποια είναι τα σχέδια τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία τηρώντας την ε, ιδιωτικότητα, την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία εμπίπτουν στο εθνικό επίπεδο, σε εθνικής, ε, στην εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιε βελτιώσει πρόσφατα. Η νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, για παράδειγμα, όπου έχουμε υποβάλει κάποιε σχετικέ ε, προτάσει, η Επίτροπο κυρία Μάλστρομ, και οι προτάσει αυτέ εξετάζονται τώρα από το Κοινοβούλιο και επίση υποβάλλουμε ορισμένες, έχουμε υποβάλει ορισμένε προτάσει όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Γιατί, όπω είπατε πολύ ορθά, είμαστε όλο και περισσότερο εξαρτημένοι ψηφιακά, άρα είναι σημαντικό να υπάρχει ελευθερία σε αυτό το ψηφιακό χώρο, αλλά με έναν υπεύθυνο χώρο. επίση να προστατεύουμε σημαντικά δικαιώματα όπω το δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα, στην ιδιωτικότητα. Άρα η προστασία των δεδομένων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και η Επιτροπή έχει υποβάλει κάποιε προτάσει που τηρούν την ισορροπία μεταξύ ελευθερία, η οποία είναι διαπραγμάτευτη, και ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το Ιντερνετ με έναν υπεύθυνο τρόπο. Ο κύριο Βότσον. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, μας έδωσε απαντήσεις για το Wikileaks. Θέλω να το ρωτήσω για κάτι για, τον οποίο, για, το, οποίο δεν έχουν, για το οποίο δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει οι πληροφορίες. Σχετικά με τα ευρωομόλογα, ε, αντιλαμβάνομαι και μοιράζω κάποιες από τις ανησυχίε που εκφράστηκαν σχετικά με την έκδοσή τους. Αλλά έχετε αναγνωρίσει την ικανότητα δανεισμού που υπάρχει σαν αποτέλεσμα της ε, ε, διαχείριση του ευρώ και επειδή ο κ. Βέτινγκ μας λέει ότι χρειάζεται 200 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια για, ενεργειακές, για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια το χρόνο για την αντιμετώπιση τη πρόκληση τη ενεργειακή ασφάλεια και τη κλιματική αλλαγή. Φιλόδο... Αυτό θα είναι κάτι το πολύ φιλόδοξο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μήπω λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτείτε την έκδοση ευρωμολόγου για τη χρηματοδότηση των υποδομών αντί για τη χρηματοδότηση της, ε, των δαπανών των κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή. Δεν ήρθα εδώ ε, για να συζητήσω μαζί σας ε, για τις wiki διαρροές. Στην, στην ομιλία μου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την έκδοση ευρωομολόγων και ομολόγων για έργα, για έργα υποδομής για να μην αυξηθεί το χρέος, διότι υπάρχει πρόβλημα υπερβολικού χρέους στην Ευρώπη, ενώ χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν μεγάλα έργα υποδομής με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως είπατε και εσείς. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει στο πρόγραμμά μας και στις προτάσεις μας για τις δημοσιονομικές προπτικές τον Ιούνιο. Θα υπάρξουν σχετικές προτάσεις, ελπίζω ότι θα ε, γίνουν δεκτές με ευρεία συνένεση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν περιορισμοί στους προπολογισμούς των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται χρηματοδότηση για ουσιαστικά αμυγό ευρωπαϊκά ε, έργα υποδομών. Ευχαριστώ. Κύριος Βεν Γίγκολτ. Okay. Uh, Mr. Uh, Romeva Iruveda. el κύριος Pero Πρόεδρε, Έχω την εντύπωση ότι αντί να μπαίνουμε στην ουσία του προβλήματος σκοτώνουμε τον ε, ταχυδρόμο. Το πρόβλημα που έδειξε, που προέκυψε από το Wikileaks ήταν το περιεχόμενο. Στο παρελθόν εσείς ο, και ο κύριος Μωρατίνος μεταξύ άλλων αρνήθηκαν ότι υπήρξε συμμετοχή των Ευρωπαίων σε μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων των ΗΠΑ. Τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Περιμένουμε λοιπόν απάντηση από πολλούς, πολλά Υπουργεία Εξωτερικών της Ένωσης και από εσά. Είναι λοιπόν βασικό να εξηγήσετε τι γίνεται ως προς το περιεχόμενο. Άλλη ερώτηση. Η εκστρατεία κατά του Julian Assange. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει το άτομο αυτό σήμερα πραγματικά είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι έκανε κάτι αναγκαίο να θέσει επιτάπητο στην αλήθεια. Και αυτό ελπίζω να το καταλάβετε και εσείς και αυτό προσδοκούμε όλοι από εσά στο Κοινοβούλιο. Εδώ ή σε μια επιτροπή που θα ενεργοποιήσουμε εκ νέου για να διαπιστώσει την αλήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επί της ουσίας, όλες οι, όλες πληροφορίες ε, που αναφέρονται αφορούν δραστηριότητες των κρατών μελών και όχι της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη μπορεί να απαντήσουν και θα απαντήσουν δίνοντας όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις γιατί είναι δημοκρατικά κράτη. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη ξεκίνησαν πρωτοβουλίε για να ε, ρίξουν φως σε κάποιε πράξει για τις οποίες ε, έγιναν, υπήρξαν καταγγελίες. Η Επιτροπή από πλευρά τη θα συμβάλλει ε, ώστε να δώσει στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη όσε περισσότερες πληροφορίε γίνεται. Για τον κύριο Ασάντζ δεν έχω τίποτα να πω. Υπάρχουν ε, ποινικέ κατηγορίε εναντίον του από ένα κράτος μέλος στη Σουηδία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που απεστάλλει από τις στις Βρετανικές αρχές, ούτε επ' αυτού έχει να πει κάτι η Επιτροπή, νομίζω ότι ενώσο δεν δικάζεται, υπάρχει η κασία, ε, υπάρχει τεκμήριο ε, Ο κ. παπα Στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πραγματικός πόλεμος δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εδώ και λίγες μέρες χιλιάδες hackers εξαπολύουν διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον των εταιριών που επιχειρούν να κατεβάσουν από το διαδίκτυο τη wikileaks ή να τη χτυπήσουν οικονομικά και να την αποκόψουν από τις δωρεές. εταιρείες όπως η mastercard η visa η paypal δέχθηκαν ηλεκτρονικές επιθέσεις τύπου ddos δηλαδή χιλιάδες υπολογιστές προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στην ίδια σελίδα υπερφορτώνοντάς την και θέτοντάς την εκτός λειτουργίας. αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό δημιουργεί γενικό πρόβλημα στις συναλλαγές των πολιτών και το ερώτημα είναι σαφές θεωρούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο ασφαλείας που να προστατεύει αυτές τις διαδικτυακές συναλλαγές των πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις. σας ευχαριστώ πολύ. δεν είστε απόλυτα προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό διατυπώσαμε κάποιες προτάσεις για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τις ε, επιθέσεις ε, από τον κυβερνοχώρο. Έχουν διατυπωθεί οι προτάσεις και λαμβάνουν υπόψη κάθε είδους τέτοιων επιθέσεων. Σχετικά με αυτές τις συγκεκριμένες στις οποίες αναφερθήκατε, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται ότι έδωσε οποιασδήποτε οδηγίες σχετικά με τις πιστοτικές κάρτες όπως είναι η Mastercard. Δεν μπορώ λοιπόν να πω τι κάνουν οι εταιρείε εξυπηρετούν ή όχι τη Wikileaks και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε και πώς, ποιες είναι οι θέσεις και των δύο πλευρών. Η κυρία Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, η δημοσίευση της διπλωματικής της, της αλληλογραφίας της, αμερικανικής διπλωματίας ε, μας έδειξε ότι υπάρχει ένα χάσμα στο σύστημα ε, αμερικανικής ασφάλειας όσον αφορά το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας. Τι συνέπειες θα έχει αυτό στο διπλωματικό επίπεδο, στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Αμερικής και ημών. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα ασφαλείας, το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, καθώς και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να παράσχουμε προστασία έναν τέτοιων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτό το οποίο συνέβη στις ΗΠΑ μπορεί να βλάψει οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σύστημα το οποίο να είναι εθαρκισμένο έναντι τέτοιου είδους επιθέσεων που θα μπορούσαν να αφορούν στον κυβερνοχώρο. Το αμερικανικό σύστημα βάσει των πληροφοριών που λάβαμε επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ωστόσο για το ευρωπαϊκό σύστημα είναι αδύνατον επίσης να εξασφαλίσουμε μια ασφάλεια 100%. Γι' αυτό συμφωνούμε ε, σε μια συνεργασία με τους Αμερικανούς φίλους μας για να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια, βεβαίως ε, σεβόμενοι τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι σημαντικό, συνεπώς, να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο βασικών αρχών πρόληψης. Λόγω των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων, αλλά θα πρέπει να τηρούμε την αρχή της σωστής ισορροπίας. Η κυρία Σονία Αλφάνο. Κύριε Πρόεδρε, όπως δείχνουν ε, οι δηλώσεις εκπροσώπων πολλών κρατών, η ερευνητική αδιαφορία, η ερευνητική μονή κατά του Ασάντς δείχνει ότι ε, προκύπτει από το ότι έδειξε στον κόσμο αυτά που έδειξε το Wikileaks με ε, η κυρία Κλίντον ζήτησε από τις Αμερικανικές πρεσβείες στη Μόσχα και τη Ρώμη πληροφορίες σχετικά με προσωπικές επενδύσεις του Μπερλουσκόν και του Πούτιν που μπορούν να θέσουν υπό αίρεση τις εξωτερικές πολιτικές των χωρών αυτών. Ε, ο, ο Μπερλουσκόνη χαρακτηρίστηκε ως εκπρόσωπος, ε, ως φερέφωνο του Πούτιν στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει μια επίθεση, αυτό προκύπτει ότι η επίθεση κατά του Ασάντζ ήταν ότι έδειξε στον κόσμο κάποιες ε, σκιές ε, στις κυβερνήσεις. Η... Η... Ο κύριος Ασάντς πρέπει να πληρώσει αν έχει κάνει κάτι δίκαια. Να ρωτήσω επίσης από την Επιτροπή να παρακολουθήσει ούτως ώστε το εργα... η ιστορία αυτή να μην χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθεί η ελευθεροτυπία και για να μην χτυπηθεί το ίντερνετ που δείχνει ότι ακόμα μια φορά είναι ένα βασικό εργαλείο προστασίας της δημοκρατίας και γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται. Ευχαριστώ. Όπως είπα νωρίτερα, δεν μπορώ να σχολιάσω επί συγκεκριμένων περιπτώσεων ή κατηγοριών ποινική ή άλλη φύση. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σάντζ, υπάρχει μια κατηγορία που έχει απαγγελθεί από την εισαγγελία τη Σουηδία που εξετάζεται τώρα από το Βρετανικό δικαστικό σύστημα. Και η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σέβονται το κράτο δικαίου θα συνεχιστεί η νόμιμη διαδικασία. Δεν μπορώ να σχολιάσω και θα πρέπει να σχολιάσω την εξέλιξη αυτή, διότι σέβομαι, σεβόμαστε και το τεκμήριο της αθωότητας και τα δικαιώματα του καθενός. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια. Για τα σχόλια που κάνατε σχετικά με το τι περιείχαν το περιεχόμενο των Wikileaks. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τα σχολιάσω. Γιατί είναι σχόλια που έχουν γραφεί από διπλωμάτες των ΗΠΑ και στέλνονται σε Πολιτικού τον είπα. Είναι δική του ευθύνη, δική του δουλειά. Δεν τα σχολιάζω. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μα θέση. Δεν είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση μας, η θέση της Ευρώπης είναι σαφής. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε τώρα σε σχόλια για συγκεκριμένες διαρροές είτε από το Wiki είτε εκτός Wiki. Ο Με κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εξακολουθούμε να χάνουμε την ουσία, τουλάχιστον νομίζω ότι στι απαντήσει σα χάνεται η ουσία. Πρώτα απ' όλα μου κάνει τεράστια εντύπωση και θέλω αν δημιουργείται και σε εσά η ίδια εντύπωση να μου το πείτε. Αυτή η απίστευτη σιωπή των ευρωπαϊκών οργάνων γύρω από την καταπίεση τη ελευθερία του λόγου. Δυστυχώ και από αυτή την αίθουσα. Όλοι οι υπερασπιστές τη ελευθερία του λόγου απουσιάζουν. Έχουν εξαφανιστεί το ερώτημα μου είναι βλέπετε μια αξιοποίηση μια χρησιμοποίηση αυτού του πράγματος για να κατασταλεί η δυνατότητα της μετάδοσης πληροφοριών. εμείς όλοι που φωνάζουμε για το δικαίωμα στο ίντερνετ των κινέζων των κουβανών και πάρα πολύ σωστά τώρα που υπάρχει μια καταστολή κυριολεκτικά αυτού του δικαιώματος τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε τι μπορείτε και πρέπει να κάνετε σαν κομισιόν. το ερώτημα δηλαδή είναι συγκεκριμένο τι θα κάνετε για να μπορεί ο πολίτης της ευρώπης να μπει στην ιστοσελίδα του wikileaks. το ουσιαστικό ερώτημα. Η ελευθερία της έκφρασης σε όλες τις μορφές της δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για τις δημοκρατικές κοινωνίες κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες ιδιωτικού, εμπορικού ή νομικού χαρακτήρα που από τη φύση τους είναι ευαίσθητες και δεν μπορούν να είναι προσιτές σε όλους. Η προστασία των δεδομένων είναι μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν κανόνες για την προστασία τους και έχουν συστήματα για, που εφαρμόζουν για την προστασία του κοινού συμφέροντος σχετικά τώρα με ε, κάποιο συγκεκριμένο άτομα. Εγώ δεν είμαι δικαστήριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώνει σχόλια για κατηγορίες που απευθύνονται κατά συγκεκριμένων ατόμων, διότι επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο και δεν μπορεί να αποφασίσει ναι ή όχι αν κάποιος είναι ένοχος. the new NATO concept Κύριε Πρόεδρε, το νέο μοντέλο του ΝΑΤΟ προϋποθέτει έναν ε, συντονισμό όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Πώς βλέπετε εσείς, ε, κύριε Πρόεδρε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια, ένας καλύτερος συντονισμός της υπεράσπισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και αυτό σχέση με το ΝΑΤΟ. Ε, τι προτίθεται να κάνει η κυρία Άστον, θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της κοινή ε, πολιτικής άμυνας. Ε, θα πρέπει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή έρευνα στο πλαίσιο αυτό του ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα. Αυτό δεν εμπίπτει βασικά στην αρμοδιότητα τη Επιτροπή. Είναι εμπίπτει στην αρμοδιότητα τη κυρίας Άστον ω ε, είπα τη εκπροσώπου. Και πράγματι αναπτύσσει αυτό το είδο ε, δράση με του βασικού μα εταίρου. Και μπορώ να σα πω, στη τελευταία συνάντηση κορυφή με τον πρόεδρο κ. Ομπάμα, ε, συζητήσαμε ακριβώ τη μορφή συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο. Γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, όχι μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά στο επίπεδο των διμερών σχέσεων με τη ΣΥΠΑ. Και πράγματι εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρέ απειλέ όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο. Ορισμένε από τι χώρε μέλη και η δική σα χώρα έγιναν αντικείμενο επιθέσεων στον κυβέρνο χώρο και αυτή είναι μια ένα σημαντικό κίνδυνο. Και έχουμε προχωρήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι ένα θέμα που οι χώρε μέλη έχουν ορισμένε ευθύνε και είπα ότι εκπρόσωπο αναπτύσσει τι προσπάθειε στην κατεύθυνση του συντονισμού, ε, ούτω ώστε να υπάρξει προστασία του κυβερνοχώρου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντέρεκ Βόγκαν. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγινε πολύ, δόθηκε πολλή δημοσιότητα σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και κάτι που προβληματίζει και απασχολεί τους ανθρώπους είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι πολλοί προβληματίζονται για το άτομο το συγκεκριμένο. Αυτό που τους προβληματίζει είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν... Καλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερους εταίρους σε αυτές τις συνομιλίες, όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών, ε, αλλά και με άλλους φορείς και οργανισμούς ανά την Ευρώπη, διότι η προστασία του κυβερνοχώρου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να συμμετάσχουν στις διαδικασίες και η τοπική και η περιφερειακή αυτοδίκηση. Γι' αυτό αυτή είναι η γραμμή που ακολουθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ε, παρακολούθησε τα γεγονότα στην Λιθουανία και στην Εστονία πριν από λίγα χρόνια ε, ε, διαρκώς δεχόμαστε επιθέσεις κατά από τον κυβερνοχώρο κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ανταποκριθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Στις 30 Σεπτεμβρίου διατυπώσαμε μια πρόταση για μια οδηγία κατά των συστημάτων ασφάλειας μετά από την ε, ανανεώνοντας την απόφαση πλαίσιο του 2005 ώστε να καταπολεμήσουμε επιθέσεις που στοχεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσιλωμένοι σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι η πρόταση οδηγίας είναι πολύ καλή, καταδικάζει και απαγορεύει ορισμένα μέσα και εργαλεία και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες αν υπάρχουν αιτήματα από, τα, από τον δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή του αιτήματο για βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργέντζο. Πρόεδρε, οι απαντήσεις που δώσετε για την υπόθεση Ασάντς και την φυλάκισή του αυτή τη στιγμή θυμίζουν λίγο δηλώσεις Πόντιου Πιλάτου. Τρεις παρατηρήσεις. Υπάρχει φούμους περσεκουτιώνης. Οι κατηγορίες είναι εξαιρετικά δύναμες. Οι ΙΠΑ ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες ζητώντα την έκδοσή του και δεν έχουν δώσει ακόμα τις νομικές αιτίε του αιτήματο αυτού. Κλείνονται τραπεζικοί λογαριασμοί. Ένας πολίτης έχει τη δυνατότητα να μην λάβει στο χώρο, στη χώρα του οικονομική υποστήριξη. Επιπλέον, οι στατιστικέ δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι υπέρ της ελευθερία στο ίντερνετ και υπέρ τη ελευθερία εν γέννη. Παρά τι ε, αμφιβολίες που δημιούργησε η πρωτοβουλία αυτή, που δεν συμμερίζομαι απόλυτα. Θέλουμε να γνωρίζουμε από τον πρόεδρο Μπαρόζο ποια είναι τα όρια και ποιο το πραγματικό θεμέλιο της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας έκφρασης. Έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό Γκουαντάναμο, ένα κίνδυνο λογοκρισίας εκ των προτέρων. Αυτές τις απαντήσεις πρέπει να δώσετε και να ελέγξετε και τις συνθήκες φυλάκισής του. Δεν, μπορεί, δεν είναι μαφιόζος για να τον έχουμε σε πλήρη απομόνωση. Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τη νομική διάσταση του θέματος χωρίς να προδικάζω βεβαίως την τελική κατάσταση. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Πρώτον, ο κύριος Ασάντς τέθηκε υποκράτηση από τις Βετανικές Αρχές βάσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης μετά από ε, ε ποινική δίωξη του κυρίου Ασάντς βάσει του ποινικού δικαίου της Σουηδίας. Αυτή ήταν η βάση πάνω στην οποία εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το, με βάση την απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, άρθρο 28, ένα άτομο που παραδίδεται μέσω του ε, εντάλματος δεν εκδίδεται σε τρίτη χώρα χωρίς τη συνένεση του κράτους που έκανε τη διαδικασία παράδοση στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο κύριος Σασάντζ κρατήθηκε τέτοια υποκράτηση στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανικές αρχές θα αποφασίσουν αν που θα αποφασίσουν αν θα τον παραδώσουν ή όχι στη Σουηδία θα πρέπει να δώσουν εκ των προτέρων τη συνένεση για την περαιτέρω έκδοσή του στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, αγαπητέ, ε, αγαπητέ κύριε Βουλευτά. Επί τη ουσία, όπω σα είπα, για την ενοχή του κύριου Ασάντ δεν μπορώ να δώσω οποιαδήποτε άποψη. Ευχαριστώ. Κύριε Λάτφορντ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Κύριε Βαρόζο, κάνατε μία δήλωση σχετικά με το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Όμω το θέμα ε, των έκδοκτων παραδόσεων δείχνει, ε, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με αυτό, ότι γύρω στα 12 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη συμμετείχαν σε αυτά τα δικήματα όπως ε, βασανιστήρια και παράνομη ε, ε, κράτηση ή μεταφορά ε, φαίνεται ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν σεβάστηκαν το άρθρο 6 της συνθήκης και τους παρακινούμε να μας πούνε την αλήθεια σχετικά με το τι έγινε και να αναλάβουν δράση βάσει του άρθρου 7, δηλαδή κυρώσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα από αυτού. Αυτό ε, εκθέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατηγορία της υποκρισίας. Τι θα κάνετε τώρα για την νομική και πολιτική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, καταχρήσεις στα πλαίσια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Ο κύριος Μπαρόζο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, εμπλακεί σε οποιοδήποτε είδο συγκάλυψη ε, παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει. Έχει καθαρό μητρό για τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν θέματα όμω που είναι ευθύνη των κρατών μελών και αυτά πρέπει να κάνουν το καθήκον του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια συνθήκη, έχουμε ευθύνε, έχουμε αρμοδιότητε, έχουμε δικαιώματα. Και θέλω να σα πω ότι η Κομισιόν έδωσε όλη τη συνεργασία που ζητήθηκε σε αυτό το Κοινοβούλιο με πλήρη διαφάνεια για τα θέματα που μόλι αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ο κύριο ευχαριστώ πρόεδρε. Και για το Wikileaks ε, που συνεχίζονται οι, δημοσίευσεις, οι δημοσιεύσεις ε, ε απόρριτων πληροφοριών και είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Ταυτόχρονα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι νόμιμη η διαδικασία με αυτά τα Wikileaks. Ταυτόχρονα στο Cyber Creek αναφέρεται ότι υφίσταται, υπάρχουν οι ε, υπέρ των επιθέσεων αυτών ή κατά και βλέπουμε εδώ ότι εδώ τώρα πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> θα κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση Κάνατε λόγο για τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτρόπου Μάλμστρομ. Υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο και κάποιες απόψεις και παρακαλώ να δοθεί σαφής απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι να δοθούν κάποιες ε, ε, λεπτομέρειες για αποφάσεις λέει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προγραμματίζει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει ε, προώθηση των ε, μεταφορών δεδομένων προς τις ΙΠΑ προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν σχεδιάζουμε καμία δράση, να αναλάβουμε δράση εναντίον του Wikileaks. Δεύτερον, όσον αφορά τις οδηγίες, τις έχουμε προτείνει και βρίσκονται προς συζήτηση και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει προτάσεις για την ε, ενίσχυση της, ε, του καθεστώτος ασφάλειας Κάποια από αυτά τα θέματα που με ρωτήσατε είναι πάρα πολύ λεπτομερή και θα προτιμούσα να σας δώσω τις πληροφορίες σε επίπεδο τεχνικών ε, πυρογνωμόνων. Ε, δεν μπορώ σε ένα λεπτό να σας τα πω όλα αυτά. Οι υπηρεσίες μου είναι στη διάθεσή σας για κάθε λεπτομέρεια που τυχόν θέλετε για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Αλλά βασικά αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με επιπτώσεις βέβαια σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα που χρησιμοποιείται χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Είναι ένα σοβαρό και σημαντικό θέμα, δεν το υποτιμώ, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφεί σχετικά με το ποιε είναι οι αρμοδιότητέ μας. Αλλά επαναλαμβάνω, ε, είμαι στη διάθεσή σας να οργανώσουμε ένα briefing ε, εντελώς πλήρες και σε τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο πρόσφατα συνέβη όσον αφορά φοροτέλος και επίθεση, επίθεση από τους hacker στην Visa, Mastercard ήθελαν να υπονομεύσουν φυσικά αυτά τα δίκτυα και να δημιουργήσουν οικονομικές απώλειες. Αυτά τα, αυτές οι επιθέσεις δημιούργησαν προβλήματα και κάποια προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα των πελατών τι απέγιναν. Αυτά τα στοιχεία ήταν ευάλωτα ή όχι. Υπάρχει κάποια δυνατότητα μέσω αυτών των ε, επιθέσεων να έχουν υποστεί κάποια ζημιά <clears throat> μόνο όταν θέλουν να αποκομίσουν χρηματοοικονομικό όφελος επιτίθενται οι hackers. Πληροφορίες, χρηματοοικονομικές και προσωπικά στοιχεία διέρευσαν και ποιος εμπλέκεται και ποιος εμπλέκεται για την αντιμετώπιση. Ποιος εμπλέκεται για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Θα ήθελα επίσης να ξέρω αν οι Αμερικανικές αρχές και οι διεθνείς αρχές εξετάζουν και διαρευνούν το θέμα. Δεν έχω άμεσες πληροφορίες ε, για τις ε, διαρροές ε, και κατά πόσον σε ποιο βαθμό εμπιστευτικά στοιχεία ιδιωτικού χαρακτήρα διέρευσαν ή όχι. Δυστυχώς λυπούμε, δεν έχω, αυτά τα ε, δεν έχω πληροφορίες, δεν έχω καμιά σχέση με αυτή την περίπτωση. Τώρα, τούτων λεχθέντων, Φυσικά αυτή η περίπτωση, αυτό το θέμα έθεσε σημαντικότατα θέματα όσον αφορά την ασφάλεια. Αληθεύει αυτό. Κάποια από αυτά τα προβλήματα ήδη τα αντιμετωπίζαμε προηγούμενα, πριν από αυτήν την περίπτωση Wikileaks. Και σα ανέφερα για τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είμαι βέβαιο και ότι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού υπήρχε και από εκεί ανησυχία, με λίματα και φροντίδα. Είμαι βέβαιο ότι γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με τη ΣΥΠΑ για να αυξηθεί η κυβερνοασφάλεια. Σεβόμενοι πάντα τι θεμελιώδει ελευθερίε διότι η ελευθερία της έκφρασης είναι φυσικά ένα, θα έλεγα, αναπαλωτρίωτο δικαίωμα για μας, ένα θεμελιώδες δικαίωμα επί του οποίου δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε. Και να δούμε και με τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία. Θα αναλυθούν λοιπόν πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουν να συγκεραστούν αυτά τα δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα ως θέματα αρχής. Σας ευχαριστώ. 21 συνάδελφοι ήταν στον κατάλογο. Μόνο 14 όμως από εσάς μπόρεσαν να παρέμβουν. Λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με τη σειρά επί του καταλόγου όπως είχε προβλεφθεί έγιναν οι παρεμβάσεις ακριβώς και ολοκληρώθηκε ο χρόνος ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Μπαρόζο, σας ευχαριστώ όλους σας συνάδελφοι για μια πάρα πολύ ζωντανή και ενθερμό συζήτηση.